σε όλες. Όπως και προηγουμένως στη συνεδρίαση των συντονιστών, θα ήθελα να σας εκφράσω τις καλύτερες ευχές μου. Ναι, Ελπίζω ότι όλοι ξεκουραστήκατε, περάσατε ωραίες διακοπές τον Αύγουστο και όλοι με μεγάλο κέφι αρχίζουμε τις εργασίες μας σε αυτή την τόσο υπεύθυνη δουλειά την οποία θα πρέπει να επιτελέσουμε. Στη συνεδρίαση των συντονιστών συζητήσαμε για το μεγάλο όγκο εργασίας τον οποίο πρέπει να φέρει σε πέραση η Επιτροπή μας. Αρχίζουμε σήμερα, πρέπει να πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 20 θέματα τα οποία είναι ακόμη εκρεμή προς ολοκλήρωση από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Η σοσιαλιστική ομάδα, όπως συζητήσαμε, θα πρέπει και προηγουμένως να εκλέξει τον συντονιστή της και θα σας αναγγείλουμε το όνομα αύριο. Η Επιτροπή μας συνεδριάζει σήμερα όλοι την ημέρα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και αύριο το πρωί την 5 3 Σεπτεμβρίου. Όπως συζητήσαμε λοιπόν και με τους συντονιστές πρέπει να δούμε ποια είναι τα κριτήρια κατανομής των εκθέσεων, που, των θεμάτων που παραμένουν εκκρεμοί όπως είπα και προηγουμένως. Σήμερα έχουμε μία αρκετά φορτωμένη ημερήσια διάξη, έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα θέματα που αφορούν και την Σουηδική Προεδρία και την παρουσίαση των προτεραιοτήτων και του προγράμματος της Σουηδικής Προεδρίας από κάποιους υπουργούς. Θα αρχίσουμε πρώτα απ' όλα από την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας έχει διανεμηθεί η ημερήσια διάταξη. Δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις αλλαγής της ημερήσιας διάταξης, άρα εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Το επόμενο σημείο. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν έχω να κάνω καμία ειδική ανακοίνωση αυτή τη στιγμή. Το μόνο που πρέπει να σας επαναλάβω είναι ότι οι συστάσεις που θα κάνουν οι συντονιστές για την κατανομή των εκθέσεων θα γίνουν αύριο το πρωί, στην αρχή της συνεδρίασης. Το επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη, είναι το πρόγραμμα εργασίας και τα επίγοντα θέματα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου. Of all pending legislative procedures has been circulated. Σας έχει κατανεμηθεί ο κατάλογος Τον έχετε στη διάθεσή σας όλοι όσοι είστε εδώ παρόντες. Η Επιτροπή μας προτίθεται να επιβάλλει πριν από το τέλος του έτους κάποια θέματα και πριν από την επόμενη συνεδρίαση οι συντονιστές και οι υπεύθυνοι των πολιτικών ομάδων θα προτείνουν τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε κατά προτεραιότητα. Για κάποιες διαδικασίες νομοθετικές, θα αλλάξει η νομική βάση εάν τεθεί σε ισχύ στην δίκη της Λισαβόνας πριν από την τελική της δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα. Αυτή είναι μια πρόταση που βασίζεται στον τρίτο πιλότνα για τα θέματα που μας απασχολούν. Η νέα νομοθετική διαδικασία επισήμως λοιπόν θα τεθεί σε ισχύ και θα ήθελα να έχουν αυτό κατά νου οι εισηγητές. Καθώς επίσης και για τα άλλα όργανα που θα συνεργάζονται στο ίδιο πνεύμα. Δηλαδή η νέα συνθήκη θα αλλάξει ορισμένες από τις υφιστάμενες νομικέ βάσεις ή θα διευρύνει το φάσμα εφαρμογή τους ή μάλιστα και θα δημιουργήσει νέες ε, νομικές βάσεις ή θα περάσει από την ομοφωνία σε ε, ενισχυμένε πλειοψηφίε. Αυτό για παράδειγμα για την ε, νόμιμη μετανάστευση και αυτές είναι οι προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας. Εν προκειμένου σε αυτές τις περιπτώσεις το έργο το οποίο ήδη έχει επιτελεστεί θα ε, είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη νέα νομοθετική εργασία. Και οι εισηγητέ θα πρέπει να διαπραγματευτούν με, τις άλλες, με τα άλλα θεσμικά όργανα γνωρίζοντα την εξέλιξη αυτή. Τέλο, η νέα συνθήκη θα ενισχύσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου σε διεθνεί διαπραγματεύσει για συμφωνίε που έχουν σχέση με αστυνομική και ε, ε συνεργασία αστυνομιών και δικαιοσύνης για την ώρα θα αναμένουμε το ε, Ιρλανδικό δημοψήφισμα, το οποίο θα ε, επηρεάσει την εξέλιξη αυτή. Όταν γίνει θα γνωρίζουμε τα πράγματα ε, περίπου σε ένα μήνα δηλαδή. Τότε στην Επιτροπή μας θα επανεξετάσουμε το πρόγραμμα εργασιών μας. Για την ώρα πάντως ζήτησα από τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι έτοιμη να μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις σας για τα θέματα αυτά. Και μου απάντησαν ότι με μεγάλη χαρά θα ενημερώσουν την παρούσα Επιτροπή σχετικά με τον ποιο τρόπο η νομική υπηρεσία μπορεί να υποστηρίξει το νομοθετικό μας έργο. Ο κύριος Καϊόλα από την νομική υπηρεσία. Η νομική υπηρεσία είναι παρούσα και είναι στη διάθεσή σας για να σας δράμει από νομικής πλευράς κατά τη διάρκεια των οργασιών σας. Όπως γνωρίζετε, η νομική υπηρεσία έχει ως κύρια αποστολή να βοηθά στην νομοθετική εργασία του τις κοινοβουλευτικέ επιτροπές κατά τη διάρκεια της, κοινοβουλίου και για οποιαδήποτε θέμα που μπορεί να τεθεί από νομικής πλευράς κατά τη διάρκεια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νομική υπηρεσία επίσης έχει ως αποστολή να προσπίζει τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εθνικές και ευρωπαϊκές δικαιωτικές αρχές. Είμαστε λοιπόν εδώ, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα νομική φύση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να το εκπροσωπήσουμε. Όπω και εσεί υπογραμμίσατε, πιθανώ η συνθήκη τη Λισαβόνα να τεθεί σε ισχύ σύντομα και σε αυτή την περίπτωση θα γίνουν σημαντικές αλλαγές στους τομείς που απασχολούν την Επιτροπή σας, ιδιαίτερος, όπως είπατε, σε θέματα που αφορούν την αστυνομική συνεργασία, την ε, συνεργασία σε θέματα ποινικού δικαίου, σε θέματα που αφορούν την συναπόφαση και θα υπάρχουν και αυξημένες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα διαπραγμάτευσης και σύναψης διεθνών συμφωνιών. Είμαστε στη διάθεσή σας σήμερα αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις αλλά και ενδεχομένως στο μέλλον είμαστε εδώ για να σας παράσχουμε την οποιαδήποτε νομική συμβουλή ή συνδρομή μας ζητήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Καγιόλα. Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο σε σχέση με τα θέματα, τα εκρεμή, τους φακέλους εκρεμής που έχουν προς εξέταση, ακόμη τους οποίους προανέφερε προηγουμένως. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις της ε, θέσης σε ισχύ της ε, Συνθήκης της Λισαβόνας σχέση με τις εργασίες της Επιτροπής μας. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Όχι. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπα και προηγουμένως, η συνεδρίαση των συντονιστών συζήτησε το θέμα των επιπτώσεων της θέση στη τη της συνθήκης της για κάποια από τα θέματα τα οποία, των οποίων η εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί από την Επιτροπή μας και θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε μια κάποια μέθοδο για να μπορέσουμε να κατανείμουμε αυτές τις εκκρεμείς εκθέσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Μποσούτλ, σύμφωνα με αυτή την ε, ε, μεθοδολογία και με την κατηγοριοποίηση των θεμάτων ανάλογα με τις επιθυμίες κάθε πολιτικής ομάδας μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή την κατανομή και όταν θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και με την ε, συνδρομή της ε, νομικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως μας εξήγησε και ο κύριος Καγιόλα, θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με τον, ανάλογα με την ε, πρέπουσα διαδικασία κάθε φάκελο χωριστά. Εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συμπληρωματικές ερωτήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, δεδομένου ότι η υπουργό Δικαιοσύνης της Σουηδίας θα έρθει στις 11. Είναι στις 11 το ραντεβού που έχουμε με την κυρία Υπουργό. Άρα διακόπτουμε στις 11 για να πιούμε καφεδάκι. Λοιπόν, 11 παρα 5 παρακαλώ να επανέλθουμε στην αίθουσα.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 So, dear colleagues, dear colleagues, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πάρτε τις θέσεις σας θα πρέπει να ξεκινήσουμε πραγματικά να αρχίσουμε τις εργασίες μας μετά από ένα σύντομο διάλειμμα. Να υποδεχθούμε φυσικά την Σουηδό Υπουργό Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Την κυρία Άσκ. Είναι τιμή μας η παρουσία της εδώ. Η κυρία Άσκ φυσικά είναι προεδρεύουσα για τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων εκτός από τα θέματα μετανάστευσης με τα οποία ασχολείται ο Υπουργός, ο συνάδελφός της Τόμπιας Μπίλστρομ τον οποίο θα έχουμε ανάμεσά μας σήμερα το απόγευμα. Η κυρία Άσκ είναι υπεύθυνη και για το θέμα της διαφάνειας των θεσμικών οργάνων. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας. Παράλληλα με τον κύριο Μπίλστρομ είναι υπεύθυνη και για την προετοιμασία του λεγόμενου προγράμματος της Στοκόλμης ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω θα διαμορφώσει μια νέα εικόνα στον τομέα της ελευθερίας, των ελευθεριών μάλλον, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης την επόμενη πενταετία. Ε, δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε ότι το θέμα αυτό είναι βασική προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο σε έφθετο χρόνο θα υποβάλει τις συστάσεις του προς το Συμβούλιο Υπουργών. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης θα είναι ε, κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό για όλους, εφόσον, όπως ελπίζουμε, μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο για τη συνθήκη της Λισαβόνας όταν αυτή τεθεί σε εφαρμογή. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προοπτικής και πριν σας δώσω το λόγο να κάνετε την παρουσίασή σας κυρία Άσκ, και ερμηνεύοντας ελπίζω το σύνολο των, μελών εδώ θα ήθελα να ζητήσω από τη Σουηδική Προεδρία να θεωρήσει ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέρος στην προετοιμασία κάποιων φιλόδοξων προγραμμάτων τα οποία βρίσκονται υπό εξέταση από το Συμβούλιο σε αυτή τη φάση θα ήθελα να τη ζητήσω να εμπλέξει περισσότερο το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στον τομέα της δικαιοσύνης. Μας ενδιαφέρει λοιπόν σαφώς να προσκληθούμε στην επόμενη συνάντηση ε, υπουργικού επίπεδου, συνάντηση κορυφής υπουργικού επίπεδου, η οποία θα γίνει στη Washington ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείε για τις δύο συνθήκες. A huge achievement and its implementation will require also the support of this parliament. So it seems to για τις δύο συνθήκες λοιπόν που θα έχουμε υπογράψει με τις Ηνωμένε Πολιτείες στον τομέα των εκδόσεων πρέπει το Κοινοβούλιο να λάβει μέρος στην επεξεργασία αυτών των συμφωνιών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Άσκα και μετά η κυρία Άσκα θα είναι στη διάθεσή σας. Θα ακούσουμε τους συναδέλφους συντονιστές πρώτα από τις πολιτικές ομάδες. Αλλά ξεκινάει η, την παρουσίασή της η κυρία Άσκ. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή στα αγγλικά και μετά όπως μου είπαν θα μιλήσω τη Σουηδική. Είναι μεγάλη χαρά, <clears throat> κανοποίηση για μένα που είμαι εδώ. Είχα έρθει την Άνοιξη εδώ για πρώτη φορά για ένα πολύ σημαντικό σεμινάριο για τα θέματα της διαφανείας. Και νομίζω ότι είναι συμβολικό το ότι η δεύτερη επαφή μας είναι πάντα στην ίδια αίθουσα. Σας περίμενα να επιστρέψετε ουσιαστικά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ε, έχουμε περιμένει και την δική σας προετοιμασία για να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αγαπητά μέλη λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντάς σας όλους όσους εξελέγησαν ή επανεξελέγησαν στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να συγχαρώ ειδικά τον κύριο Λόπες Αγκουιλάρ ε, γιατί έγινε πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Η Σουηδική Προεδρία θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία μαζί σας. Θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες στον τομέα της δικαιοσύνης και των δημοσίων ελευθεριών. Ε, τώρα μιλάμε για ένα τομέα ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, πάρα πολύ ευρύσος. εκ τούτου ελπίζω να με συγχωρήσετε γιατί θα θέσω τις βασικές γραμμές της πολιτικής μας και μετά θα δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις στις απορίες σας. Ο συνάδελφος Μπίστρον το απόγευμα θα δώσει απαντήσεις σε θέματα όπως η πολιτική χορήγηση θεωρήσεων καταπολέμησης της ε, παράνομης μετανάστευσης και χορήγησης ασύλου. Έχουμε λοιπόν στον τομέα μου πολλά προβλήματα, την σωματεμπορία, την λαθρεμπορία, την εμπορία ναρκωτικών ουσιών και έχουμε και νέου τύπου παραβατικές συμπεριφορές και εγκλήματα, εγκλήματα τα οποία τελούνται μέσω του ίντερνετ και τα λοιπά. Θα πρέπει να υπάρξει <clears throat> συνεργασία για την καταπολέμηση των απειλών αυτών. Έχει αυξηθεί η συνεργασία αυτή, υπάρχει σήμερα, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να συνεργαστούμε στενότερα σε θέματα τήρησης τάξης και σε θέματα δικαιοσύνης. Το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη και όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και εκτός Ευρώπης είναι κάτι το οποίο αγνοεί τα εθνικά σύνορα. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι τα εσωτερικά ή διοικητικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά στην καταπολέμηση της, του οργανωμένου εγκλήματος. Δυστυχώς είναι πολύ σημαντικό το οργανωμένο έγκλημα σήμερα και όλοι περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει με τα μέτρα τα οποία λαμβάνει για την καταπολέμηση αυτής, της, αυτού του φαινομένου. τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε πρέπει φυσικά να βελτιώσουν ε, την αίσθηση ασφάλειας χωρίς να παραβιάζουν ε, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τον ιδιωτικό χώρο των πολιτών. Η προοπτική των πολιτών, επαναλαμβάνω, είναι η βάση επί της οποίας εδράζουμε τις προσπάθειές μας. Σε επίπεδο βέβαια θεσμικό, συνταγματικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε μια ανασφαλή κατάσταση και θα ήθελα το ταχύτερο δυνατό να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία της Λισαβόνας. Η συνθήκη της Λισαβόνας περιλαμβάνει βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής μας στον τομέα της δικαιοσύνης, ενισχύει φυσικά και τον δικό σας ρόλο, και θα μας επιτρέψει αυτό να συνεργαστούμε καλύτερα και στενότερα στο μέλλον ελπίζω. Η επεξεργασία του προγράμματος της Στοκχόλμης, το οποίο συνιστά θα έλεγα το επόμενο πενταετές πρόγραμμα δράσης μας, είναι ο πιο βασικός στόχος της Σοηδικής Προεδρίας, λέει η κυρία Άσκ. Στόχος της Σουηδικής Κυβέρνησης είναι να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι ταυτόχρονα φιλόδοξο, ρεαλιστικό και ε, δίκαιο θα έλεγα για όλους. Να δείχνουμε μέσω του προγράμματος αυτού την μεγάλη σημασία που έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της επίτευξης των πολιτικών στόχων που έχουμε θέσει. Μακροπρόθεσμα σημαντικό επίσης πρέπει να είναι το πρόγραμμα αυτό, γιατί θα θέλαμε να ενισχύσουμε ακόμα τη συνεργασία μας, η οποία να μην περιορίζεται χρονικά από την πενταετή αυτή χρονική περίοδο. Και θα πρέπει να είναι και ισόρροπο το πρόγραμμα αυτό, ισόρροπο και δίκαιο, γιατί το πρόγραμμα θα πρέπει να αντισταθμίζει τα μέτρα αυτά τα οποία είναι κατασταλτικής φύσεως, με μέτρα τα οποία θα προστατεύσουν την ατομική θα αξιοπρέπεια και τις βασικές ελευθερίες και δικαιώματα των πολιτών. Βάση λοιπόν, θεμέλιο του προγράμματος της Στοκόλμης είναι ένα σύνολο μέτρων τα οποία αντικατοπτρίζουν τις φιλοδοξίες που έχουμε και τις προσπάθειες να ισορροπήσουμε τα κατασταλτικά μέτρα από τη μία με την προστασία των δικαιωμάτων από την άλλη. Κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν κάναμε όσο έπρεπε. Σύνεπως, το σημείο εκκίνησης της προσπάθειάς μας είναι η ανακοίνωση του μηνός Ιουνίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την πρώτη φορά που το συζητήσαμε αυτό ε, ήταν σε επίπεδο υπουργικό, ανεπίσημη συνάντηση τον μήνα Ιούλιο και ο, ο πρόεδρός σας, ο κύριος Λόπες Αγουιλάρη, ήταν παρόν και αυτό το εκτιμήσαμε όλοι. Βέβαια όλα έγιναν την τελευταία στιγμή και δεν μπορέσαμε να προγραμματίσουμε σωστά τη συνεργασία μας. Παρόλα αυτά θα έλεγα εκτιμήσαμε το γεγονός ότι μπόρεσε να είναι παρόν σε μια τέτοια πρώτη φάση. Βασικά ε, ε, υπάρχει μια κάποια συνένεση για την ε, βασική γραμμή που θα ακολουθήσει η ανακοίνωσή μας. Πολλοί συνάδελφοι υπουργοί υπογράμμισαν την σημασία της προοπτικής αυτής η οποία προέρχεται από την βάση όπως είπα από τον πολίτη. Στο μέλλον η συνεργασία μας θα πρέπει να βασίζεται σε ορισμένα μέτρα τα οποία θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την συνεχή προσπάθεια την οποία κάνουμε. Ένας άλλος τομέας στον οποίο πρέπει να πάρουμε μέτρα είναι η ανάγκη ανάλυσης της, των νομοθετικών μέτρων τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και αξιολόγησης των νομοθετικών αυτών μέσων. Έτσι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της νομοθετικής δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την συμβατότητα των μέτρων μεταξύ τους και την ευκολία στην πρόσβαση του κοινού και των ειδικών που θα μπορούν να διαβουλεύονται και να εφαρμόζουν την νομοθεσία που έχει ήδη υιοθετηθεί. Όλα αυτά λοιπόν θα θέλαμε να τροφοδοτήσουμε με όλα αυτά να τροφοδοτήσουμε το πρόγραμμα της Στοκόλμης. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και δυσκολίες για, την, για τον αμοιβαίο σεβασμό των διαφορετικών συστημάτων των νομικών τα οποία ισχύουν σήμερα. Πάντως ε, πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ μας, η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση, πρέπει να υπάρξουν μέτρα εμπιστοσύνης παράλληλα μέσω ανταλλαγών, πληροφόρησης, κατάρτισης. Όλα αυτά θα βελτιώσουν την μεταξύ μας κατανόηση και συνεργασία. Ε, συζητήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος Εράσμους για εισαγγελείς και δικαστές. στα όργανα τα οποία έρχονται σε επαφή με τους πολίτες, η αμοιβαία γνώση των νομικών συστημάτων είναι σχετικά περιορισμένη. Και αν δεν κατανοεί κάποιος κάτι σε βάθος, δεν είναι ε, σε κατάσταση να αποδώσει την δικαιοσύνη όταν αυτή απαιτείται επιτόπου. Συνεπώς λοιπόν μπορούμε με πρακτικά μέτρα να βελτιώσουμε το κλίμα εμπιστοσύνης. Ένα άλλο μέτρο για τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης είναι να συμφωνήσουμε σε ελάχιστα στάνταρς για διαφορετικές περιπτώσεις παραβατικότητας. Δηλαδή, ελπίζω να πετύχουμε κάποιους κοινούς στόχους εναρμόνισης ε, της δράσης μας και θα πρέπει επίσης μέσω πρόθεσμα να προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε και κάποιες υποχρεώσεις στα πλαίσια του προγράμματος της Στοχόλμης. Να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου και ότι θα προστατεύονται τα δικαιώματα των προσώπων. Πολλοί θα έχετε ακούσει για ανθρώπους που ταξιδεύουν πολύ στην Ευρώπη και που έρχονται σε επαφή με άλλα δικαιικά συστήματα τα οποία δεν γνωρίζουν καλά, δεν τα κατανοούν, δεν γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Εδώ μπορούμε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία. Για την συνεργασία στην πράξη. Εκεί διάφορες αντιπροσωπείες στην ε, συνάντηση της Στοκχόλμης τόνισαν ότι εδώ μπορεί να παίξει έναν ενισχυμένο ρόλο η Ευρωπόλ μέσα στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Συνεργασίας, αλλά και όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο διεθνές. Και σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε διάφορα είδη εγκλημάτων, πιλωτικούς τομείς που θα θεωρήσει ότι έχουν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την ανάγκη μελέτης συστημάτων αντιμετώπισης τους. Για παράδειγμα, σωματεμπορία, γενετής εκμετάλλευση παιδιών, εγκλήματα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαφθορά και ούτω καθεξής. Εκεί χρειάζεται η συνεργασία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορέσει να είναι μια τέτοια συνεργασία αποτελεσματική. Στις συζητήσεις που έγιναν στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, διάφοροι συνάδελφοί μου τόνισαν και πόσο σημαντικές είναι οι εξωτερικές σχέσεις. Τα εξωτερικά επομένως σήμερα, σύνορα της ε, που δεν είναι βεβαίω σύνορα τα οποία αποτρέπουν τους εγκληματίες από το να δραστηριοποιούνται και εδώ πρέπει τα πράγματα αυτά να ληφθούν υπόψη περισσότερο στο μέλλον. Από τις συζητήσεις η εντύπωσή μου που διεξήχθησαν δηλαδή σε αυτό το άτυπο συμβούλιο στη Στοκόλμη είναι ότι συνολικά συμφωνούμε επί των βασικών γραμμών της μελλοντική συνεργασίας και η Προεδρία καλείται τώρα να συλλέξει τις διάφορες αυτές απόψεις και να φροντίσει ώστε να περάσουν στο τελικό σχέδιο του προγράμματος το οποίο θα υποβληθεί και θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης τον ε, Σεπτέμβριο. Και ελπίζω ότι θα συνεχιστούν οι επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένω με ενδιαφέρον το ε, ψήφισμα το οποίο θα υποβάλλεται και θα ψηφίσετε τον Σεπτέμβριο. Ο γραμματέας του Υπουργείου μου, Μάρκους Κράνα, για θέματα ε, μετανάστευσης έχει το καθήκον ε, να ε, διευθύνει τις σχετικές συζητήσεις. Έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι θα προσέλθει στις δικές σας κοινοβουλευτικές επιτροπές δημοσίων ελευθεριών και δικαιοσύνης και ο υπουργό κ. Μπίλστρομ θα έλθει επίσης αργότερα το φθινόπωρο για να συζητήσει μαζί σας. Θα επανέλθουμε σε συζητήσεις μαζί σας Νοέμβριο. Άλλο μέγα θέμα είναι η διαφάνεια. Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών και καλύτερης κατανόησης του έργου μας. Η διαφάνεια είναι σημαντικό θέμα και για εμάς τους Σουηδούς και γνωρίζουμε ότι και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο αποτελεί προτεραιότητα. Ο κανονισμός περί διαφάνειας που ισχύει τώρα εγκρίθηκε την άνοιξη του 2001 στην τελευταία ε, Σουηδική Προεδρία πριν από την ε, τωρινή. Και ορισμένοι εξημών ήσασταν ήδη τότε ε, στο Κοινοβουλίο και είχατε αναμειχθεί στην προσπάθεια αυτή. Νομίζω ότι ο κανονισμός αυτός αποδίδει. Έχει περιλάβει πολύ ισορροπημένες λύσεις που φροντίζουν και για το κοινό καλό, αλλά και για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών. Ταυτόχρονα πρέπει να καταστεί σαφέστερη η νομοθεσία και σε ορισμένα σημεία πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες που προκύπτουν από την εφαρμογή στην πράξη. Ελπίζουμε το φετινό φθινόπωρο να, μπορούμε να, επιτύχουμε, να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό θα χρειαστεί βέβαια σκληρή δουλειά, αλλά και διάθεση για παραχωρήσεις από όλες τις πλευρές. Τα τεχνικά θέματα συζητούνται τώρα στο Συμβούλιο. Υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί. Όμως αποκρισταλώνεται σιγά, σιγά σιγά η θέση αυτή του Συμβουλίου. Και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και ποιε πρωτοβουλίε θα αναλάβει το Κοινοβούλιο. Από πλευρά Σουηδική Προεδρία ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την ίδια δέσμευση όπως το 2001, ώστε να καταλήξουμε σε μια λύση που να εγγυάται καλύτερη και αποτελεσματικότερη νομοθεσία σε ό,τι αφορά θέματα διαφάνειας. Είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι είναι απαραίτητο να αναζητηθούν κοινέ λύσεις για τα διάφορα προβλήματα. Η Ευρώπη χωρίς σύνορα ασφαλώς και γίνεται και αντικείμενο κατάχρησης από πλευρά του οργανωμένου εγκλήματος. Τα εσωτερικά σύνορα στην Ευρώπη δεν επιτρέπεται να εμποδίζουν και εμάς του ίδιους στην προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Χρειαζόμαστε άρα ικανοποιητική, αποτελεσματική συνεργασία αστυνομιών, ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Η Ευρωπόλ για μας είναι σημαντικό εργαλείο για την διευκόλυνση της συνεργασίας αυτής τη ειδικότητα της συνεργασίας στην Ευρώπη. Η Ευρωπόλη, η οποία πρόκειται να εορτάσει και την δεκαετία από τις ίδρυσεώς τη και που έχει το σημαντικό καθήκον να ενισχύει την συνεργασία για την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματο. Θα γίνει σύντομα στην Χάγη ειδική συνάντηση με συμμετοχή και της Ευρωπόλ για την καλύτερη οργάνωσή της. Και βεβαίως ε, θα προσκληθεί και ο πρόεδρος σας. Νομίζω μάλιστα έχει ήδη ε, γίνει η πρόσκληση. Όπου θα συζητηθεί εκεί ο ρόλος της Ευρωπόλ και οι περαιτέρω εργασίες. Εάν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματική συνεργασία επέκεινα των συνόρων, πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και ανταλλαγή πληροφοριών, αναλόγως με τις ανάγκες που προκύπτουν. Οι εθνικές αστυνομικές αρχές έχουν ορισμένες φορές την ανάγκη να κάνουν τέτοιες ανταλλαγές πληροφοριών. Εμείς επιθυμούμε να ενισχυθεί και η συνεργασία στο τομέα της δικαιοσύνης. Με βελτιστοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών, ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη ασφάλεια υπερόλων. Υπάρχουν και ορισμένες πληροφορίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από κοινού. Έχουμε και ορισμένες προδιαγραφές για την διατήρηση των πληροφοριών αυτών, οι οποίες δεν πρέπει να ε, αποθηκεύονται και να διατηρούνται επάπειρον. Θα γίνουν προτάσεις από τη Σουηδική Προεδρία και για αυτή τη μελλοντική ανταλλαγή πληροφοριών. Βέβαια, ο σκοπός είναι πάντοτε η καταπολέμηση βαριών εγκλημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες και για την καθημερινή ζωή, για την στάση ορισμένων πολιτών σε θέματα θρησκευτικά ή πολιτικά. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια ασφαλέστερη Ευρώπη, ταυτόχρονα να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα αποτελεσματικά, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσουμε την προσωπική σφαίρα δεν είναι το δίλημα ή το τρίλημα αυτό άλυτο. Μπορεί να ε, δοθεί λύση. Οι πληροφορίες που ε, θα πρέπει να ανταλλάσσονται θα πρέπει να είναι υψηλή ποιότητα, μεγάλη αξιοπιστία. Αυτό ισχύει και για τα αποδεικτικά μέσα, όπω για παράδειγμα δακτυλικά αποτυπώματα. Η τεχνολογία έχει, που χρησιμοποιούν δηλαδή οι διοκτικές αρχές έχουν, έχει βελτιωθεί πολύ. Η προσπάθεια δηλαδή να συνδεθεί ένα συγκεκριμένο δράστη με ένα συγκεκριμένο έγκλημα είναι σημαντική, έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση. Έχουμε και προτάσεις που γίνονται από σουηδικής πλευράς για την τεχνολογία της ε, δίωξης, ιατροδικαστικά και άλλα. Και πρόκειται εδώ για μια προσπάθεια να ε, θεσπιστούν κοινέ προδιαγραφές που να επιτρέπουν την χρήση των πληροφοριών αυτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θέλουμε η πρωτοβουλία αυτή να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του έτους και θα παρακαλέσουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει το δυνατόν συντομότερο την γνωμοδότησή του ώστε να μπορέσει να ληφθεί υπόψη στις διαβουλεύσεις. Ορισμένοι θεωρούν ότι τα θέματα αυτά είναι περισσότερο τεχνικά, όπως και η όλη η ιατροδικαστική τεχνολογία. Εγώ θεωρώ πάντως ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους πολίτες, διότι όλοι κατανοούν πόσο σημαντικό είναι, για παράδειγμα, όπως του σιδηροδρόμους, είναι σημαντικό όλες οι σιδηροδρομικές γραμμές σε όλη την Ευρώπη να έχουν το ίδιο εύρο, το ίδιο πλάτος για να μπορούν να κυκλοφορούν οι σύρμοι με ευκολία. Το ίδιο κατανοείται βεβαίως ότι πρέπει να ισχύει και για θέματα τεχνολογίας αλλά και συλλογή των πληροφοριών. Και αυτό ενδιαφέρει τους περισσότερους συμπολίτες μας. Τέτοια θέματα ακούγονται ακόμα και σε τηλεοπτικές αστυνομικές σειρές και είναι προφανές πόσο πολύ απασχολούν τους πολίτες. Ο θεμέλιος λίθος για, την, για το δικαστική συνεργασία είναι αυτή η απαραίτητη εμπιστοσύνη μεταξύ των εθνικών αρχών, αλλά και η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στα μέτρα τα οποία προτιθέμεθα να εγκρίνουμε. Οι χώρες μέλη και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται οι μεν τις δε, αναγνωρίζοντας δηλαδή τις κρίσεις των άλλων και θα πρέπει να διασφαλίζουμε ελάχιστες προδιαγραφές στους πολίτες, ελάχιστες προστασίες δηλαδή. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι θα διαθέτουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα σε οποιαδήποτε χώρα ε, βρίσκονται ε, από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα μπορούν δηλαδή να πληροφορηθούν εφόσον ε, τους απαγγελθεί κατηγορία σε μια γλώσσα την οποία είναι κατανοητή σε αυτούς περί τίνος πρόκειται αυτό άλλωστε είναι και αποτελεί και τη βάση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από πλευρά Σουηδική προεδρία για τα διαδικαστικά δικαιώματα, για τα δικονομικά δικαιώματα των πολιτών. Δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα να υπάρξει μια απόφαση πλαίσιο για τα θέματα αυτά. Και γνωρίζω ότι και πολλά εθνικά κοινοβούλια συμμερίζονται την άποψή μας αυτή. Έχω συζητήσει το θέμα με όλους σχεδόν τους υπουργού δικαιοσύνης και θεωρώ ότι έχουν βελτιωθεί οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε πρόοδο εν προκειμένου. Και αν δεν μπορέσουμε τελικά να επιτελέσουμε πρόοδο, τότε αυτό σημαίνει ότι μπλοκάρουμε, ότι στην ουσία υπονομεύουμε την περαιτέρω συνεργασία μας. Υπονομεύουμε ολόκληρη τη συνεργασία στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι χώρες μέλη θα πρέπει να συντάξουν ένα είδος οδικού χάρτη για το πώς θα εφαρμοστούν σταδιακά τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα με τρόπο ώστε και ο πολίτης να βλέπει ότι υπάρχει μια προστιθέμενη αξία σε αυτά και το πρώτο βήμα θα έπρεπε να είναι ένας κοινός μηχανισμός για μεταφράσεις και διερμηνία σε περιπτώσεις όπου ασκούνται διώξεις. Οι πολίτες αναμένουν τις πρωτοβουλίες αυτές από εμάς και αναμένουν και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την διασφάλιση των δικαιωμάτων ουδήποτε προσώπου κατηγορείται για κάποιο αδίκημα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή αντιμετώπιση του. Συχνά οι σχετικέ εμπειρίες είναι τραυματικές. Τραυματικές για ολόκληρη τη ζωή του θυγωμένου. Και είναι πολύ δυνότερη κατάσταση όταν αυτό συμβαίνει σε μια ξένη χώρα όπου το θυγόμενο πρόσωπο δεν γνωρίζει την ενόμη τάξη, δεν γνωρίζει τις διαδικασίες, δεν γνωρίζει ποια δικαιώματα έχει ή ποιες υποχρώσεις. Πολύ συχνά λοιπόν αισθάνεται απόλυτα εκτεθειμένος ο άνθρωπος αυτός και είναι ε, βαρύτατες οι τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να αποκομίσει. Η ελευθερία διακίνησης εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει επίση ότι αυξάνεται και ο αριθμός των προσώπων εκείνων που ενδέχεται να τους απαγγελθεί κατηγορία για κάποιο αδίκημα στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν, η κατηγορία αυτή εφόσον απαγγελθεί θα πρέπει να είναι σε μια γλώσσα κατανοητή για αυτούς. Πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν επί μιας στρατηγικής που να υποστηρίζει περισσότερο και τα θύματα εγκληματικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, μια εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των θυμάτων και των δραστών ή ενδεχομένως δραστών, ώστε να μην υπάρχει διάκριση σε βάση ε, φίλου θρησκείας, ε, ηλικίας ή εντοχμένης αναπηρίας. Και το θύμα λοιπόν πρέπει να υποστηρίζεται και να ε, του εξασφαλίζεται μια αποζημίωση για την ζημία την οποία υπέστη <clears throat> λόγω ενός αδικήματος ε, για ενός εγκλήματος βίας. Και εν προκειμένου αναμένω την επικοδομητική σας συνεργασία για την υποστήριξη, όπως είπα, και των θυμάτων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Μιλώντας για ασφάλεια δικαίου, είναι σημαντικό να πω ότι και αυτός που έχει υποστεί ε, το αδίκημα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει στις δικαστικές διαδικασίες, αλλά και να είναι και ενήμερος. Υπάρχουν πολλοί τομείς όπου οι χώρες μέλη οφείλουν να συνεργαστούν, κυρίως βέβαια στην καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, κυρίως ε, αναφέρομαι εδώ στην σώματεμπορία, εκεί χρειαζόμαστε ακόμα αυστηρότερα μέτρα, ιδιαίτερα για την προστασία των παιδιών, για παράδειγμα κατά της παιδικής πορνογραφίας ή και άλλων ε, γενετήσεων πονογραφίας η μέρα να μην ανοίξετε την εφημερίδα και να δείτε ότι κάτι τέτοιο πάλι έχει συμβεί. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αναλυφθεί ο αγώνας αυτός. Ο αγώνας κατά της σωματεμπορίας έχει ύψιστη προτεραιότητα για την Σουηδική Προεδρία. Η σωματεμπορία, κυρίως σε βάρος παιδιών ή γυναικών, αποκρουστικό αδίκημα το οποίο χρειάζεται απαραίτητα διεθνή συνεργασία για να αντιμετωπιστεί. Το φθινόπωρο θα διαπραγματευτούμε σχέδια προτάσεων του Συμβουλίου που να μας δώσουν τους απαραίτητους μηχανισμούς, αλλά όπως είπα, η συνεργασία μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αρκεί. Χρειάζεται συνεργασία και με τις τρίτες χώρες, και τις χώρες προέλευσης των ε, προσώπων αυτών. Όπως είπα, έχουμε αποδώσει ύψιστη προτεραιότητα στο θέμα της σωματεμπορίας και στις επαφές μας με τρίτες χώρες. Θα ε, οργανώσουμε από τις 19 20 Οκτωβρίου ε, διεθνή διάσκεψη με συμμετοχή αρμοδίων και από τρίτες χώρες. Θεωρούμε ότι είναι καλός ο τρόπος αυτός για ανταλλαγή απόψεων, για συλλογή πληροφοριών και να ε, κάνουμε και ένα oriented paper. Θα υποστηρίξουμε και διμερείς ε, συνεργασίες για την ε, διασυνοριακή καταπολέμηση του εκδήματος. Βεβαίως προσκαλείται και το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στην διάσκεψη αυτή του Οκτωβρίου. Είναι σημαντικό επίσης να εγκύψουμε στο θέμα της ασφάλειας των παιδιών, διότι η τεχνολογικές εξελίξεις βαδίζουν με γοργό ρυθμό και αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Το ίντερνετ δεν γνωρίζει σύνορα και έχει διευκολύνει πολύ την διάδοση της παιδικής πορνογραφίας καθώς και των πρακτικών γενετήσεω κατάχρησης παιδιών. Εδώ πρέπει να λάβουμε αυστηρά μέτρα για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε τους δράστες. Ήδη τον Ιούνιο η Κομισιόν έχει εκδώσει σχετικό έγγραφο και είναι σημαντικό το θέμα. Στο θέμα αυτό προωθούμε τις διαπραγματεύσεις, για παράδειγμα και του σεξουαλικού τουρισμού και το λεγόμενο grooming, όταν δηλαδή ενήλικοι προσπαθούν μέσω του ίντερνετ να έλθουν σε επαφή με νεαρά παιδιά με ε, σκοπούς γενετήσιας εκμετάλλευσής τους. Εδώ χρειάζεται ενημέρωση των παιδιών. Παλαιότερα φροντίζαμε να ε, προειδοποιούμε τα παιδιά να μην ακολουθήσουν ποτέ κάποιον ενήλικο ο οποίος μπορεί να του φαίνονταν περίεργο. Τώρα δεν φτάνει αυτό να βγουν απλώ στον δρόμο. Τώρα υπάρχει ο κίνδυνο του ίντερνετ που έρχεται μέσα στα σπίτια. Η Σουηδική Προεδρία θα προωθήσει και θα υποστηρίξει και άλλε μεθόδου συνεργασία στον αγώνα κατά της γενετήσιας κατάχρησης η εκμετάλλευση των παιδιών, για παράδειγμα εθελοντική συνεργασία και στον οικονομικό τομέα. Για παράδειγμα, μπορούμε να φανταστούμε ότι τράπεζες ή εταιρείες πιστοτικών καρτών μπορούν να διακόψουν τις online πληρωμές σε τέτοιες περιπτώσεις, σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της γενετήσιας εκμετάλλευσης των παιδιών. Και όταν θα μπορούν να συνεργαστούν οι αρχές δικαιοσύνης, θα χρειαστεί να αναλυθούν και άλλες πρωτοβουλίες, τις οποίες εμείς θα προωθήσουμε. Τελειώνω σιγά σιγά. Θέλω να θυμίσω ακόμη ότι με 15 χώρες μέλη έχουμε υποβάλει μια πρωτοβουλία που συζητείται τώρα στο Συμβούλιο Υπουργών για την ποινική δίωξη και την μεταφορά της ποινική δίωξης σε άλλη χώρα. Εφόσον δηλαδή η ποινική δίωξη μεταφέρεται από μία χώρα μέλος σε άλλη, τότε βέβαια πρέπει να υπάρχουν και κοινοί κανόνες οι οποίοι να διέπουν την δίωξη αυτή. Βέβαια, περιοριζόμαστε στους πιο σημαντικούς τομείς, ώστε να διεξάγονται και με αποτελεσματικό τρόπο οι δικαστικές διαδικασίες. Αυτό είναι σημαντικό και για τους δικαστές και για τα θύματα των αδικημάτων χρειαζόμαστε και ένα κοινό πλαίσιο για αυτές τις μεταφορές των ποινικών διώξεων. Και επειδή βλέπουμε ότι αυξάνονται διασυνοριακά τα εγκλήματα, συχνά υπάρχει ανάγκη δίωξη ταυτόχρονα σε πολλές χώρες. Εκεί χρειαζόμαστε κοινά κριτήρια. Ήδη έχουμε τη συνεργασία των αστυνομιών, την συνεργασία των δικαστικών αρχών για την επιβολή κατασταλτικών μέτρων. Εν προκειμένου αναφέρω και το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως. Βέβαια, προσπάθειες πρέπει να γίνονται και για την υποστήριξη των θυμάτων και αυτά τα θύματα δηλαδή πρέπει να ενημερώνονται για μια ενδεχόμενη μεταφορά της ποινική διώξεως. Αυτό ισχύει και για την, ε, ειδικότερα για την σωματεμπορία. Οι ανακρίσεις θα πρέπει να γίνονται συγκεντρωτικά σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά τους, γιατί για την ώρα είναι πολύ κατακαιρματισμένες οι ανακριτικές διαδικασίες. Ελπίζω ότι και αυτό το έγγραφο θα μπορέσει να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, Αυτά είναι λίγα από τα σημαντικότερα θέματα που ε, έχω επί της τραπέζης μου τώρα στην Σουηδική Προεδρία. Θα ήθελα εν τέλει να εκφράσω την ελπίδα μου ότι θα συνεχίσω με την θετική συνεργασία με την ε, Επιτροπή σας τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και αναμένω τα σχόλια και τις ενδεχόμενες ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ, Υπουργέ, για την προσεκτική παρουσίαση των προτεραιοτήτων και των λεπτομεριών της πολιτικής της Προεδρίας. Είναι καιρός να δώσουμε το λόγο στα μέλη που έχουν ζητήσει τον λόγο. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Ο Ντιάς Ντεμέρα πρώτα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ξέρετε ότι οι τρία λεπτά μπορείτε να μιλήσετε. Υπάρχει περιορισμός χρόνου για να μπορέσουμε να ακούσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό μελών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την δυνατότητα να μιλήσω εκ μέρους του ΕΛΚ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που μας εκθέσετε με τόσες λεπτομέρειες το πρόγραμμά σας. Το ΕΛΚ συμμερίζεται εξ ολοκλήρου όλες τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Αργότερα θα ασχοληθούμε με τα θέματα της μετανάστευσης και βεβαίως της σωματεμπορία που συνδέονται μεταξύ τους. Θα ήθελα να σας πω ότι όντως η Στοκχόλμη ως ε, επέκταση του προγράμματος της ε, ΧΑΗ θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να λύσουμε τα θέματα που μας απασχολούν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα ή πέντε συγκεκριμένα θέματα και να σας υποβάλω ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, κυρία Υπουργέ, σε σχέση με τη Europol. Θα θέλαμε να ακούσουμε αν αναλάβετε τη δέσμευση, κυρία Υπουργέ, να είναι διακυβερνητική οργάνωση η Ευρωπόλ για να γίνει πραγματικά μία από τις περίφημες agencies της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και όπου όλοι οι υπάλληλοι θα είναι Ευρωπαίοι. Πράγμα το οποίο θα την βοηθήσει να ξεπεράσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει την κρίση εμπιστοσύνη που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Δεύτερη προτεραιότητα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Υπουργέ, και εσεί αναφερθήκατε ακροθυγός σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα περισσότερε λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, η Σουηδική Προεδρία να λάβει δερμεύσει για την ε, ανταλλαγή των μητρώων ε, ε, αν υπάρχει πρόβλημα στον ποινικό μητρό κάπου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε θέματα αστυνομικής συνεργασίας και συνεργασίας ε, δικαστικής. Τρίτον, θα θέλαμε δέσμευση εκ μέρου κυρία Υπουργέ, για θέματα ε, καλύτερου συντονισμού για τα θέματα της ε, δίωξης των τρομοκρατών. Έχουμε την Europol, έχουμε τον συντονιστή, ο οποίος θα έρθει να μας επισκέφθει σε θέματα τρομοκρατίας, ο οποίος θα μας επισκέφθει μετά. Έχουμε ειδικέ υπηρεσίες των κρατών μελών. Θα θέλαμε να αναλάβετε εσείς τη δέσμευση, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων αυτών των οργάνων. Ο συντονισμός απορρέει από την εξειδίκευση. Δεν ε, δίδουμε πληροφορίες σε αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν να τις χειριστούν με τον κατάλληλο τρόπο και δεν έχουν τη γνώση. Θα θέλαμε λοιπόν συντονισμό εκ μέρους σας. Επίσης θα θέλαμε ε, να υπάρχει ενίσχυση της Eurojust δέσμευση επίσης για την καταπολέμηση των παραχαρακτών του ευρώ για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα το κοινό μας ευρωπαϊκό νόμισμα. Και τελικά κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το οποίο και εσείς ε, τονίσατε την ε, καταπολέμηση του εγκλήματος σε όλες τις ε, μορφές του και κυρίως την καταπολέμηση των, ε, της παιδεραστίας. Πολλές ερωτήσεις σας έκανα και ξέρω ότι έχετε λίγο χρόνο. Αφήνω λοιπόν το χρόνο και σε άλλους συναδέλφους να μιλήσουν. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις των Σας ευχαριστώ κυρία Ντίσε Δεμέρα. Εκ μέρους των σοσιαλιστών το λόγο έχει η κυρία Μπόσκουτ. Δύο λεπτά παρακαλώ κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω την Ολλανδική. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Ελπίζω να μπορέσω να περιοριστώ στα λεπτά τα οποία τα μου ορίσατε. Θα ήθελα να θέσω ορισμένε ερωτήσεις ε, για έναν τομέα στον οποίο δεν σταθήκατε ιδιαίτερα. Ε, είναι το θέμα ίσως που αφορά περισσότερο τους, ε, το Συμβούλιο Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά αναφέρομαι στην οδηγία για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες από τη Σουηδική προσδοκία για την συγκεκριμένη οδηγία και διαρωτώ με τι σκοπεύει να κάνει η Σουηδική Προεδρία και πότε μπορούμε εμείς να αναμένουμε συγκεκριμένα μέτρα προτάσεις από πλευράς των Σουηδών για την καταπολέμηση του ρατσισμού θυμίζω ότι μετά από την αποτυχημένη συνάντηση κορυφής των Ηνωμένων Εθνών πολλές προσδοκίες διαψεύστησαν. Η Σουηδία είναι μια χώρα η οποία έχει στρέψει θα έλεγα την προσοχή της στην καταπολέμηση του ρατσισμού. Σκοπεύεται ίσως να οργανώσετε μια συνάντηση κορυφής για την καταπολέμηση του ρατσισμού κάτι το οποίο θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει την κατάσταση γιατί επαναλαμβάνονται τα φαινόμενα στην Ευρώπη τα οποία μας κάνουν να ανησυχούμε σε καθημερινή βάση. Η... Το λόγο τώρα έχει η επόμενη πολιτική ομάδα, η κυρία Πλάσκαρτ, τρία λεπτά. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό, λέει η κυρία Πλάσκαρτ, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και θα ήθελα να περιοριστώ σε μία παρατήρηση μόνο. Αναφερθήκατε σε ένα κλίμα απογοήτευσης σχετικά με τα διαδικαστικά γύρω από τις, ε, από δικαστικές διαδικασίες. Και είπατε ότι θα προσπαθήσετε σε πρακτικό επίπεδο να βρείτε κάποιες ε, λύσεις, πρώτες λύσεις για να ξεκινήσει μια συζήτηση. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος ε, Ασφάλειας και Ελευθερίας είναι ένας χώρος ο οποίος σε πολιτικό επίπεδο δεν έχει κάνει τα απαιτούμενα βήματα. Και όταν τα βήματα αυτά γίνονται, τα ίδια τα συστήματα, τα διαδικαστικά στις διάφορες χώρες δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ευρωπαϊκό ένταλμα σαν παράδειγμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, αλλά διαπράττονται πάρα πολλά λάθη και υπάρχει απογοήτευση σχετικά από την, κρίση του, από την χρήση του συστήματος αυτού. Για τη μεταφορά ενός κρατουμένου σαν παράδειγμα από τη μία χώρα στην άλλη. Οι διαδικασίες είναι πάρα πολύ περίπλοκες και είναι περίπλοκες όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς λοιπόν τι θα γίνει, θα ξεκινήσει πραγματικά ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό από το 2011. Οι διαδικασίες μεταφοράς ορισμένων δικαστικών ρυθμίσεων, αποφάσεων και νομικών προτάσεων και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις, συγχύσεις και δυσκολίες. Εν πάση περιπτώσει εγώ δεν είμαι κατά των μέτρων τα οποία ανακοινώνεται, αλλά μήπως τελικά υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν επιθυμούν να εφαρμοστούν ε, θέματα, που, θέματα, αποφάσεις μάλλον που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς μπορείτε να ξεπεράσετε τους δισταγμούς και ε, τις αντιρρήσεις των κρατών μελών, οι οποίες εκφράζονται κυρίως μέσω των παρατεταμένων διαδικαστικών ε, ε, καθυστερήσεων. Νομίζω ότι σε επίπεδο διαδικαστικό πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και πολύ γρήγορα, γιατί αλλιώς το οικοδόμημα το οποίο προσπαθούμε να στήσουμε θα κινδυνεύσει. Επαναλαμβάνω για τη μεταφορά των κρατουμένων, φυλακισμένων ή κρατουμένων. Ε, υπάρχουν προβλήματα διαδικαστικά και το πρόβλημα παραμένει χένον και θα παραμείνει έτσι τουλάχιστον μέχρι το 2011. Ο κύριος Άλμπερτ για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ για, την, για αυτά τα οποία είπατε για την καλύτερη και στενότερη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πράγματι θα πρέπει να προστατευθούν και να ενισχυθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα πρέπει επίσης να προστατευθούν και τα ατομικά δεδομένα. Μέχρι τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Το πρόγραμμά σας περιλαμβάνει αρκετά συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών, την διαδικτύωση τραπεζών δεδομένων και τη συγκεκριμένη μεταφορά ε, δεδομένων. Η συγκεκριμένη με ερώτηση τώρα είναι για τα δεδομένα SWIFT καθώς και PMR προς τις Ενωμένες Πολιτείες. Κατά πόσο αυτά αποτελούν τμήμα του προγράμματος της Στοκχόλμης. Αυτό έχει ενδιαφέρον νομίζω. Και από την άλλη μεριά εμείς οι πράσινοι βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη και προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και κυρίως της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αλλά εδώ δεν βλέπουμε να είναι πολύ ξεκάθαρες οι προσπάθειες σας. Ιδίως για τον τρίτο πυλώνα. Μήπως θα ήταν δυνατό εδώ να γίνει μια ανανέωση της απόφασης πλαίσιο για την προστασία αυτή και να περιληφθεί η προσπάθεια αυτή στην, στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης και τι γίνεται και με τις επιπτώσεις στα προγράμματα προβλέπεται αξιολόγηση. Τι γίνεται όμως με τις συνέπειες αυτής της αξιολόγησης. Θα ήταν σωστό να σημειωθεί πιο συγκεκριμένα πώς αξιολογούνται τα μέτρα και στη βάση ποιων κριτηρίων τροποποιούνται μετά τα μέτρα ή ενδεχομένως αποσύρονται κάποια μέτρα. Μέτρα τα οποία ελήφθησαν για παράδειγμα τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα της συνεργασίας αστυνομιών δικαιοσύνης, αλλά όπου αποδείχτηκε εκ των υστέρων ότι ήταν δυσανάλογα βαριά τα μέτρα αυτά σε σχέση με την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Εάν θα υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένη αξιολόγηση και υποθέτω ότι η Σουηδική Προεδρία μπορεί εδώ να δραστηριοποιηθεί πιο συγκεκριμένα. Κάτι που με ενδιαφέρει εμένα επίσης ιδιαίτερα και που θα πρέπει να περιληφθεί πιο ξεκάθαρα στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ότι αυτά τα πράγματα, η αξιολόγηση δηλαδή των υφιστάμενων μέτρων, θα πρέπει να γίνει πριν από την λήψη νέων μέτρων. Και εδώ θα θέλαμε λοιπόν να υπάρξει ε, κάπως μεγαλύτερη σαφήνεια. Σας ευχαριστώ. Θα, δώσω, δώσω το λόγο ευθύς αμέσως στον κύριο Ταβάρες της Ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς. Αλλά πρώτα θέλω να πω ότι σηκώθηκαν τόσο πολλά χέρια που θα πρέπει ε, να περιορίσουμε τον χρόνο ε, αγορεύσεώς σας. Άρα παρακαλώ μην σηκώσετε άλλα χέρια ώστε ε, να μπορέσουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις σε διαδοχικούς γύρους. Πάντως ακόμα θα ακούσουμε τώρα σε αυτό το γύρο τον κύριο Ταβάρες για τρία λεπτά της ΓουΕ και μετά θα δώσω το λόγο στην Υπουργό παρακαλώντας την να μην υπερβεί τα πέντε λεπτά περίπου. Αλλά πρώτα εσείς κύριε Ταβάρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και την διευκρινή σας. Θα ήθελα αρχίζοντας να κάνω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτα αφορά το SWIFT θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση της ε, Σουηδικής Προεδρίας σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα στο SWIFT. Εμεί θα έχουμε μία συνάντηση για αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σας άποψη, η άποψη Προεδρίας δηλαδή, σχέση με αυτό το θέμα. Για τη Europol τώρα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση της ε, Σουηδικής Προεδρίας για τον δημοκρατικό έλεγχο στην Ευρωπόλ, στα πλαίσια των συζητήσεων που γίνεται για το μέλλον της Ευρωπόλ. Τώρα, όσον αφορά τη σωματεμπορία, κυρία Υπουργέ, είπατε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα αυτό της σωματεμπορίας. Θα ήθελα να μου πείτε, υπάρχουν κάποια κριτήρια, κάποια minimum κριτήρια χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την συνεργασία με τρίτες χώρες ή πρόκειται για συνεργασία ε, γενικότερη ή συνεργασία πιο συγκεκριμένη. Τελικά, τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω δύο πιο γενικού περιεχομένου ε, κρίσεις, παρατηρήσεις. Πρώτη, αφορά κάτι το οποίο νομίζω ότι άκουσα το οποίο είπατε. Δηλαδή, μιλήσατε όχι μόνο για διαφάνεια των εγγράφων αλλά και απλούστευση, απλότητα των εγγράφων αυτών, καλύτερη κατανόηση. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό της ε, σωστής ενημέρωσης, της ε, κατανοητής ενημέρωσης προς τους πολίτες είναι καθήκον μας. Είπαμε πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει, και το είπαμε όλες οι πολιτικές μας εδώ, να έχουμε διαφάνεια παντού, αλλά δεν επαρκεί. Διότι δεν έχουν όλοι οι πολίτες τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα του περιεχομένου κάποιων δημοσίων εγγράφων. Θα πρέπει λοιπόν η απλούστευση των εγγράφων αυτών να συνοδεύει και τη διαφάνεια. Ένα άλλο γενικό θέμα αφορά, όπως είπατε κυρία Υπουργέ, την ε, ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ε, δικαιωμάτων των πολιτών. Νομίζω ότι δεν έχουμε απόλυτη ισορροπία μεταξύ ισορροπίας και δικαιωμάτων των πολιτών. Έχουμε πρώτα απ' όλα με τα, ε, στα δικαιώματα των πολιτών έχουμε αρχές και η ασφάλεια είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν μπορούμε τα δικαιώματα λοιπόν των πολιτών να τα σεβόμαστε στο περίπου ή να τα τηρούμε στο περίπου. Θα πρέπει λοιπόν να τραβήξουμε προς τη μεριά των δικαιωμάτων, να επιτύχουμε καλύτερη ισορροπία για να έχουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα σφάλμα ε, δομικό αν θέλετε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να υπάρχει επανεξισορρόπηση των δύο αυτών των. Σας ευχαριστώ. Σας δίνω το λόγο κυρία Υπουργέ για να απαντήσετε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων και μετά θα ανοίξουμε δεύτερο γύρο. Δύο λεπτά ο καθένας στη διαθεσή του. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και θα πρέπει και πάλι να δώσουμε χρόνο στην Υπουργό να απαντήσει. Ε, ε, Synpunkter och frågor. Jag ska vara väldigt kortfattad för att försöka σας ευχαριστώ πολύ και πρόεδρε. Θα προσπαθήσω, κατά το δυνατόν, να είμαι σύντομη και να απαντήσω σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Θα αρχίσω με το SWIFT και τις σχετικές συζητήσεις. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Χρειαζόμαστε τη συμφωνία αυτή με τις Ενωμένες Πολιτείες στον τομέα αυτό. Ο, ο λόγος για την ανταλλαγή και χρήση αυτών των πληροφοριών είναι βέβαια η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μία από τις πιο αποτελεσματικές δυνατότητες πλήξης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας είναι να κλείσουν οι στρόφικες των χρηματοδοτήσεων. Είναι σημαντικές οι πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει κανείς με τον τρόπο αυτό. Ταυτόχρονα, ε, εάν υπάρξει, αν επιθυμούμε να υπάρξει συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών με οποιονδήποτε. Άλλωστε πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός ώστε και οι πληροφορίες να είναι οι σωστές, αυτές που συλλέγονται δηλαδή, αλλά και ταυτόχρονα να, γίνεται, να είναι ασφαλής η χρήση τους. Στην προκείμενη περίπτωση έχουμε και εμείς ιδιαίτερο ενδιαφέρον να υπάρξει ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο για την ε, συλλογή τέτοιων πληροφοριών να είναι σαφώ οριοθετημένο το πλαίσιο. Υπάρχουν πληροφορίε που διαθέτουν οι Ηνωμένε Πολιτείε και που μπορούμε, μπορεί να μα φανούν και σε εμά χρήσιμε για την καταπολέμηση Τρομοκρατία στην Ευρώπη. Βεβαίω και οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται να λαμβάνουν πληροφορίε από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και θα ήταν παράξενο εάν εμεί δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε μαζί του, Αλλά πάντως η <clears throat> συμφωνία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και περιορισμένη. Είναι πάντως σωστό ότι γίνονται οι ε, συζητήσεις αυτές γιατί είναι περίπλοκο το θέμα. Άλλο σημαντικό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και που διαπιστώνω τώρα ότι δεν το εξήγησα πολύ, η Ευρωπόλη είναι σημαντικό όργανο, σημειοτομής αν θέλετε, πολλών συνεργασιών. Η βάση είναι η διεθνή συνεργασία. Και άλλωστε δεν θέλει κανείς να αφαιρέσει την ευθύνη από τις χώρες μέλη. Αλλά η Ευρωπόλ μπορεί να είναι ένα καλό σημείο τομής, όπως είπα, ένα σημείο συλλογής, συγκέντρωσης ε, των πληροφοριών, όπου όμως μπορούν να ε, διαπιστώσουν οι ε, αρμόδιοι και τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά για το λόγο αυτό η Ευρωπόλ θα πρέπει να μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικότερα. Είναι λοιπόν καλό που υπάρχουν οι νέοι κανόνες για την Ευρωπόλ. Γνωρίζετε όμως ότι οι νέοι θεσμικοί κανόνες που συζητούνται, η νέα ε, ηγεσία που συζητείται, απετέλεσαν και τους λόγους για τους οποίους συνεκάλεσα τους υπουργούς σε έκτακτη ε, σύνοδο με παρουσία της Ευρωπόλη για να δούμε ποια πράγματα μπορούμε να βελτιώσουμε στην συνεργασία μεταξύ Ευρωπόλ και χωρών μελών. Νομίζω ότι μπορούμε πράγματι να το επιτύχουμε αυτό, να επιτύχουμε μια καλύτερη συνεργασία. Ακούστηκε και ερώτηση για τα ποινικά μητρώα. Οι αστυνομικές οργανώσεις, αστυνομικές αρχές έχουν από καιρού ε, συνεργασία είτε με το τηλέφωνο είτε με το φαξ Νομίζω οι αστυνομικές αρχές είναι και εκείνες ε, οι αρχές στις χώρες μέλη που ανταλλάσσουν και τα περισσότερα φαξ, αν και ίσως τώρα έχουν περάσει και σε πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Πάντως αυτό που απασχολεί είναι και ο εξυγχρονισμός της τεχνολογίας, ώστε να μπορούν να δρουν και να αντιδρούν ταχύτερα. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή απαραίτητα το να αυξηθεί ο όγκο των συλλεγόμενων πληροφοριών. Αυτό που ενδιαφέρει είναι μια απογραφειοκρατικοποίηση, μια απορρίθμιση ε, και νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει τους περισσότερου. Υπάρχουν και τομείς όπου συζητήσαμε εάν ίσω χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίες. Και αυτό ο δρόμος είναι σημαντικός για την Σουηδική Προεδρία. Δηλαδή να είναι σημαντικέ, να είναι ε, συγκεκριμένες οι πληροφορίες και να αποδίδουν μια προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι σημαντικό για την Σουηδική Προεδρία. Ο Ευρωπαίος εντεταλμένος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων διάβασε και αυτό στην ανακοίνωση της Επιτροπής και ο ίδιος θεωρεί ότι η πρόταση είναι καλή, ότι αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτά δεν είχαν συζητηθεί επαρκώς προηγουμένως. Εδώ λοιπόν μπορεί πραγματικά να υπάρξει μια σημαντική διαφορά. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω είναι η παλαιά διάκριση όταν υπάρχει δηλαδή ε, κάποια αρμοδιότητα άλλου υπουργού δεν είναι ε, ε, αυτή είναι, είναι άλλη αρμοδιότητα άλλη υπουργού ε, όπως είπα για την καταπολέμηση ωστόσο της τρομοκρατίας. Εκεί έχουμε ένα τομέα, την ριζοσπαστικοποίηση δηλαδή, που ε, πρέπει να μας απασχολήσει. Σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν τόποι όπου διάφοροι άνθρωποι, νέοι κυρίως, δραστηριοποιούνται, ενδεχομένως επειδή αισθάνονται αποκλεισμένοι, αισθάνονται ότι είναι θύματα διακρίσεων, για παράδειγμα είναι δύσκολο να βρει δουλειά, ε, θεωρεί ότι δεν τον σέβονται παρκώς. Ε, η καταπολέμηση του εγκλήματος λοιπόν είναι η μία πλευρά. Αλλά και αυτή η άλλη πλευρά, δηλαδή αντιμετώπιση των διακρίσεων, αντιμετώπιση των ρατσιστικών διαθέσεων, είναι και αυτό σημαντικό. Όμως, όπως είπα, η συγκεκριμένη οδηγία ε, υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου Υπουργού και γι' αυτό ε, δεν ε, έχω άμεση απάντηση για το θέμα. Θα ολοκληρώσω εδώ και θα επανέλθω. final Λοιπόν, δεύτερος γύρος, τελικός γύρος, δύο λεπτά ο καθένας. Έχω πραγματικά μεγάλες προσδοκίες από τη Σουηδική Προεδρία και διάβασα και τις προτάσεις σας για το πρόγραμμα της Στοχόλμης και είδα ότι συγκεντρώνετε την προσοχή σας στον ίδιο τον πολίτη, στο άτομο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και είναι και μια ριζοσπαστική τομή θα έλεγα σε σχέση με το παρελθόν. Μέχρι τώρα τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου θα έλεγα έχουν υπονομευθεί από τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Φυσικά δεν, είμαι απόλυτα, δεν είναι απόλυτα καθησυχιστικά αυτά τα οποία μας λέτε. Γιατί έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά μέτρα τα οποία περιορίζουν σαφέστατα τα δικαιώματα των πολιτών. Και λέτε ότι ήταν απαραίτητα γιατί μας παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Σας πιστεύω, θέλω να σας πιστέψω, αλλά παρόλα αυτά που είναι οι αποδείξεις. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2008 περιμένουμε μία απάντηση για το ψήφισμά μας για τους προσωπικούς κωδικούς επιβατών, τα PNRs. Θέλουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν τα μεγαλύτερα επίπεδα ασφαλείας και θέλουμε να μας δώσετε μία απάντηση επιτέλους, γιατί το θέμα έχει αρχίσει και γίνεται όλο και περισσότερο ε, απίστευτο. Σχετικά με τη διαφάνεια, φυσικά και η Σουηδία έχει μία μακρά παράδοση στον τομέα της ε, διαφάνειας και της πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα. Και γι' αυτό οι υποσχέσεις σας ε, ε, είναι καλοδεχούμενες. Βέβαια θέλω να θέσω ορισμένε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, ερωτήσεις. Θα επιτρέψετε άμεση και πλήρη πρόσβαση ε, στις εργασίες της νομικής υπηρεσίας στην περίπτωση της υπόθεσης SWIFT. Θα δώσετε πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία αφορούν τις σφαιρικές διαπραγματεύσεις για το ΆΚΤΑ που δίνει ε, ιδιαίτερες δυνατότητες στους μεθοριακούς φορούς να ε, ψάχνουν και να ερευνούν τις ε, αποσκευές μας αλλά και τα λάπτοπς και τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και τι γίνεται επίσης με τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει γύρω από τις παράνομες μεταφορές κρατουμένων από τη CIA. Τελειώνω πρόεδρε. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι αξιολογήσεις οι οποίες έγιναν και στη δική μου χώρα δείχνουν ότι τα πράγματα είναι απαράδεκτα και οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες της χώρας μου έχουν καταρρεύσει και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, συνέχισε την ίδια πρακτική. Γι' αυτό λοιπόν οι αξιολογήσεις τις οποίες εσείς μας υπόσχεστε να είναι πιο αποτελεσματικές. Μωράες δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστρέψω στον πυρήνα θα έλεγα της παρουσίασής σας. Βέβαια σε λίγα λεπτά είναι δύσκολο να μιλήσετε μόνο συνολικά για όλα τα θέματα, αλλά το οργανωμένο έγκλημα και το ερώτημα ακριβώς το οποίο έθεσε και ο Ντεμέρα είναι κατά πόσον είναι αποτελεσματική η Ευρωπόλ. Εμείς το συζητάμε αυτό στο Κοινοβούλιο και εμείς πιστεύουμε ότι από το 2010 και μετά θα πρέπει πράγματι να αλλάξει ο χαρακτήρας της Europol. Εφόσον γίνει λοιπόν αποτελεσματική η Europol για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της σώματεμπορίας, τότε θα έλεγα ότι η κλίμακα του οργανωμένου εγκλήματος είναι τόσο μεγάλη που Ευρωπόλ όσο και αν βελτιωθεί θα παραμείνει μικρή. Συνεπώς λοιπόν η επιμονή σας στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και σωστότερης ενημέρωσης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και υπάρχουν πάρα πολλά και φιλόδοξα προγράμματα όπως η ανταλλαγή ιατροδικαστικών στοιχείων. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα πάρα πολύ προσεκτικά και η ανταλλαγή στοιχείων DNA και άλλων ιδιωτικών στοιχείων είναι κάτι το πάρα πολύ ευαίσθητο και γι' αυτό τι μέτρα προστασίας της, του ιδιωτικού χώρου θα ληφθούν στο συγκεκριμένο τομέα. Ξέρω ότι και τα παραδείγματα τα οποία μας δώσατε δείχνουν μια κάποια κατεύθυνση, αλλά θέλω περισσότερες λεπτομέρειες. Και όπως είπε και η κυρία Χένης Πλάσκαρτ, η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης δεν είναι η καλύτερη δυνατή και βλέπουμε ότι δεν είμαστε σε θέση εμείς να αξιολογήσουμε σωστά τα μέτρα και την εφαρμογή των μέτρων τα οποία έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε να τα αξιολογήσουμε σωστά και γι' αυτό από τη μία θα πρέπει να δούμε πώς πηγαίνουν τα πράγματα και αν πηγαίνουν αποτελεσματικά όπως τα θέλαμε, αν η Ευρωπόλ σαν παράδειγμα δουλεύει με ικανοποιητικό τρόπο και από την άλλη θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι νέες φιλόδοξες προτάσεις και πώς μπορούμε να τις περάσουμε. Η ε, κυρία Χιμένε, χίλια δύο λεπτά. κυρία ε, Υπουργέ, θα ήθελα να συγχαρώ για την παρέμβασή σας. Θα ήθελα να σας πω, όπως ήδη γνωρίζετε, ότι οι τρομοκρατικές πράξεις ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και μπορούν να πλήξουν όλη την επικράτεια της Ευρώπης. Ξέρετε ότι πρόσφατα στη χώρα μας, στην Ισπανία, έγιναν πολλές ε, τρομοκρατικές ε, επιθέσεις. Ε, στην ε, Μαγιόρκα απέτυχε μία τρομοκρατική επίθεση στο Μπούργκας Είναι ένα από τα κύρια θέματα που μας απασχολούν στην Ισπανία, όπως σας απασχολούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για μας τους Ισπανούς είναι προτεραιότητα. Διάβασα το πρόγραμμά σας και χαίρομαι που μεταξύ των προτεραιοτήτων συμπεριλάβατε και την συνεργασία σε θέματα δίωξη των τρομοκρατών. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει με την ε, ε, υιοθέτηση αποτρεπτικών μέτρων, ώστε οι φανατικοί τρομοκράτες να σταματήσουν να ενεργούν. Ακούγοντάς σας, ε, να μιλάτε με ζωηρό ενδιαφέρον υπέρ των ε, θυμάτων, θα μιλήσω και για τα δικαιώματα των θυμάτων. Σας ερωτώ, η Σουηδική Προεδρία θα εκδώσει κοινοτική νομοθεσία για να εναρμονιστούν οι εθνικές νομοθεσίες. Σήμερα είναι πάρα πολύ διαφορετικές σε θέματα ε, αρρωγής των θυμάτων της ε, ε τρομοκρατίας με ηθικά και άλλα υλικά μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν να σας προσφέρω σε τέτοιου είδους ενέργειες που θα καταβάλλετε την δική μας υποστήριξη. Εάν θέλετε μπορείτε να έρθετε σε επαφή με μένα με τους επόμενους μήνες της Σουηδικής Προεδρίας για να συνεργαστούμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εναρμονίσουμε αυτά τα μέτρα. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριο Στράσερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Υπουργό και την κυβέρνησή της για το πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που μας παρουσίασε και θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερως διότι εκπώνησε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεπερνά το εξάμεινο της ε, Σουηδικής Προεδρίας. Θα ήθελα να υποβάλω τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, η αστυνομική συνεργασία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι μας είπατε ότι δεν υπάρχουν πλέον σύνορα για τους πολίτες, αλλά δεν υπάρχουν και για τους εγκληματίες πλέον. Τα σύνορα παρόλα αυτά υπάρχουν για τους αστυνόμους και πολλές φορές θα πρέπει σε αυτή την Ευρώπη της πρόοδου να ενισχυθεί η Ευρωπόλ. Και θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά τα οποία είπε η συνάλφος Ισπανή. Χρειαζόμαστε να έχουμε μια Ευρωπολ δυνατή. Θα πρέπει να της δώσουμε νέες αρμοδιότητες για να, μπορεί, να μπορεί να εργάζεται επιτόπου, άμεσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πιο γρήγορη και καλή ενημέρωση μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να εμπνευστούμε από διάφορες ομάδες συνεργασίας οι οποίες έχουν λειτουργήσει πολύ σωστά. Επίσης, τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει κάτι να κάνει η Ευρώπη περισσότερο για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των εξωτερικών της σύνορες. Επίσης, θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά τα οποία Σπανός συνάδελφος, θα πρέπει να ενισχύσουμε τον συντονισμό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της στρατηγικής που θα υιοθετήσουμε στα πλαίσια του προγράμματος της Στοκχόλμης έγιναν κάποιες προτάσεις από την ε, Υπουργό την Αυστρία και θα ήθελα και εσείς ε, αυτές τις ε, προτάσεις να τις συνεχίσετε. κυρία Βέμπερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Έχω μία ερώτηση σας υποβάλλω. Είπατε τη διάρκεια της σας ότι υπάρχει μία απόφαση πλαίσιο για την ποινικέ διαδικασίε και τη μεταφορά και θα θέλετε να υπάρξει απόφαση μέχρι το τέλο του χρόνου. Γιατί δεν υπάρχει και απόφαση πλαίσιο ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα δικαιοδοτικά σε τέτοιου είδους θέματα. Δεδομένου ότι πρόκειται για το ίδιο πλαίσιο. Όταν υπάρχει πρόβλημα δικαιοδοτικών οργάνων θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Μιλήσατε για το τέλος του χρόνου, αλλά υπάρχουν ε, πάρα πολλές μεγάλες διαφορές ε, όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της πρότασης πλαισίου. Υπάρχουν θέματα τα οποία ρυθμίζονται, αλλά συγχρόνως υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες περιπτώσεις. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί μεταξύ αυτών των δύο αποφάσεων πλαίσιο λοιπόν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Ευχαριστώ. Η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε πόσο ανοιχτή είναι σε πολλά θέματα της εργασία η Σουηδική Προεδρία και ο στόχος μας ε, να υπάρξει ε, καλή συνεργασία με εσάς ε, Νομίζω ότι θα επιτευχθεί. Υπάρχει μεγάλη βούλη συνεργασίας, απλώς θα πρέπει να αποσαφινιστούν και κάποια πράγματα. Αυτό το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερος όταν ακούω το Συμβούλιο, είναι σε κάποιες επιχειρήσεις η προσπάθεια μη πρόσβαση σε κάποια σημαντικά έγγραφα. Υπάρχουν φάκελοι, θέματα που αφορούν διεθνείς υποθέσεις, οι οποίες παραμένουν ως απόρριτοι Και συμφωνώ με αυτά που είπε επί του θέμα της κυρία Ίτβελτ. Μπορείτε εσείς ε, τέτοιου είδους πρακτικές να τις αποτρέψετε ή να τις μειώσετε. Μπορείτε να κάνετε κάτι στο Συμβούλιο ώστε να τονιστεί περισσότερο το άνοιγμα, η πρόσβαση κάποιων στοιχείων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάλμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό Δικαιοσύνης για τον χρόνο που μας αφιερώνει. Ήδη μπορέσαμε στη Στοκχόλμη να την συναντήσουμε και να μιλήσουμε μαζί της. Σήμερα μας εξήγησε το πρόγραμμά της. Κυρία Υπουργέ, μας ε, μιλήσατε για τα χρησιμοποίηση δεδομένων DNA. Που έχουν πια ε, αποκτήσει αποδεικτική αρχή στις <clears throat> δικαστικέ διαδικασίες είτε για την καταδίκη είτε για την αθώωση. Τώρα όμως υπάρχει η συμφωνία του ΠΡΙΜ που κατέδειξε ότι είναι διαφορετικές οι ε, διαδικασίες στις χώρες μέλη για την συλλογή των δεδομένων DNA ώστε υπάρχει διαφορά και στη στατιστική αξιολόγησή τους και στην αποδεικτική τους αξία. Θα έπρεπε λοιπόν εν προκειμένου να υπάρξουν κοινέ προδιαγραφέ σε όλη την Ευρώπη, εφόσον πρόκειται να γίνουν ανταλλαγέ δεδομένων DNA μεταξύ των χωρών μελών. Άλλο θέμα τώρα. Εάν ποτέ το σκεφτήκατε ή εάν ενδεχομένω έχει κάποια σημασία μέσα στα πλαίσια τη της Λισαβόνα ε, συνθήκης ε, της Λισαβόνας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μυστικών υπηρεσιών. Υποθέτω ότι σε κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο υπάρχει ένα όργανο το οποίο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών. Ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει για το ΣΥΤΣΕΝ. Δεν γνωρίζουμε ε, οι διάφορες αυτές οι υπηρεσίες τι πράττουν. Στο κοινοβουλευτικό επίπεδο το γνωρίζουμε δηλαδή. Μιλήσατε και για την Ευρωπόλ εφόσον δώσετε επιχειρησιακές δυνατότητες στην Ευρωπόλ, μήπως τότε θα πρέπει να αρθεί η ασυλία των υπαλλήλων της Ευρωπόλ. Επίσης, η Σουηδική Προεδρία, τώρα μετά από τις ευρωεκλογές, έχει σκεφτεί με κάποιο τρόπο πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν κάποιες αναζωπυρώσεις ακροδεξιών ή εθνικιστικών τάσεων ε, στην ε, Ευρώπη. Χωρίς μικρόφωνο, μιλητής. Mike, Mike, please. Sorry. Under the European arrest warrant, will it... Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, μπορεί ε, να απελαθεί κάποιος από μια χώρα όταν έχει διαπράξει κάτι ε, το οποίο δεν είναι όμως, ε, δεν θεωρείται εν πάση περιπτώσει παράνομο στην χώρα προς την οποία ε, έχει απελαθεί. Μιλήσατε επίσης για τα προβλήματα συγχρονισμού των νομικών συστημάτων. Ξέρετε ότι η Ουαλία έχει ειδικά συστήματα. Τι θα κάνετε γι' αυτά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την λεπτομερή παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Σουηδικής Προεδρίας. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που ε, συντάχθηκε μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό κλίμα θα περιλάβει τις προσπάθειες όχι βέβαια μόνο των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όλου του κόσμου. Ε, Το ΑΕΠ σε όλες τις χώρες του κόσμου. Πέφτει, οι τράπεζες πτωχεύουν, ο κόσμος χάνει τις δουλειές του. Αυτό αναγκαστικά θα οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας και άρα ε, θα ε, δημιουργήσει ένα κλίμα πιο ευνοϊκό για πλήσιμο του χρήματος, για ε, προσπάθειες φοροδιαφυγής, για διαφθορά. Άρα πάλι ο αριθμός των οικονομικών εγκλημάτων θα αυξηθεί και οι σχετικές δίκες θα είναι πιο πολύ άριθμες. Στις διάφορες ωστόσο χώρες μέλη της Ένωσης βλέπουμε το κοινό να έχει σχετικά χαμηλή, περιορισμένη εμπιστοσύνη απέναντι στους ε, δικαστές και άλλες δικαστικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτού του πενταετούς ε, προγράμματος Στοχόλμης. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το οικονομικό έγκλημα. Ποια είναι τα πρόσθετα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και στους δικαστές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Υπουργό να της ευχηθώ ότι καλύτερο για ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα. Επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας υπογραμμίσατε την επιθυμία σας να υπάρξει στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη στον τομέα της Τζάι. Και αναφερθήκατε στο θέμα της σώματεμπορίας, στο θέμα της άσκησης βίας και μέσω της πορνογραφίας και του σεξουαλικού τουρισμού στους ε, νεότερους στα παιδιά. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο ε, σας απασχολεί ήδη και εδώ θα έλεγα θεωρώ δεδομένη την ευαισθησία σας, είναι το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών. Μας είπατε ήδη ότι υπάρχει μια επιβλητική ποσότητα θα έλεγα πληροφόρησης η οποία κυκλοφορεί ανάμεσα στα κράτη-μέλη αλλά με εντελώς ακατάλληλο τρόπο σε σχέση με την ευθετότητα του χρόνου και την ενημέρωσή τους των στοιχείων τα οποία ανταλλάσσονται. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ και το θέμα της ανταλλαγής και αμοιβαίας ενημέρωσης σχετικά με τα ποινικά μητρώα, ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για πορνογραφία και μάλιστα παιδική πορνογραφία γιατί στον τομέα αυτό υπάρχει μια σαφέστατη υψηλή ε, δυνατότητα επανάληψης του συγκεκριμένου εγκλήματος και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η πρόληψη. Ένα ερώτημα λοιπόν. Θα ήθελα να μάθω εάν η Σουηδική Προεδρία έχει την επιθυμία να κάνει προσπάθειες στα θέματα των ανηλίκων στο μέλλον. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ανηλίκων που έχουν πέσει θύματα απαγωγής και έχουν γίνει θύματα εκμετάλλευσης. Ξέρετε ότι υπάρχουν επίσης πάρα πολλά παιδιά παιδιά Ευρωπαίων πολιτών ή διαφορετικών εθνικοτήτων που μετά από το διαζύγιο ε, των γονιών τους ή στην ουσία είτε μέσω απαγωγών βρίσκονται σε άλλη χώρα είτε αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα λόγω ακριβώς της έλλειψης επικοινωνίας ε, μεταξύ των δικαστικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Αναφέρομαι στο τμήμα, στο του προγράμματος της Στοκόλμης που ασχολείται με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια ανακοίνωση και έκανε ένα ερωτηματολόγιο και θα ήθελαν το 88% αυτών που έδωσαν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς αυτό δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανησυχίες τις οποίες έχετε εσείς και στη συμπερίληψη του συγκεκριμένου θέματος στο πρόγραμμα της Στοχόλμης. Βλέπετε συγκεκριμένα μέτρα μέχρι το τέλος της Προεδρίας σας στα πλαίσια της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ή τι θα θέλατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ Αλφάνο. Ευχαριστώ και εγώ την Υπουργό Δικαιοσύνη της Σουηδίας για την παρουσία της εδώ. Πάντα στο θέμα της δικαιοσύνης. Ξέρετε ότι είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό για μια χώρα ιδιαίτερα στην Ιταλία. Γι' αυτό ακριβώς έχουν υπάρξει συγκεκριμένοι νόμοι στη χώρα μου μέσω των οποίων τροποποιήθηκε το ίδιο το Σύνταγμα. Το άρθρο 3, σαν παράδειγμα του συντάγματος, λέει ότι οι πολίτες της Ιταλίας είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Μέσω όμως ενός απλού νόμου δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο, διότι υπάρχουν διακρίσεις τελικά ανάμεσα στους Ιταλούς πολίτες. Η ομάδα των φιλελευθέρων έχει κάνει, θα έλεγα, κάποια διαβήματα και έχει προτείνει να γίνει μια συζήτηση σε σχέση με τον νόμο αυτό, ο οποίος είναι γνωστός ως νόμος Αλφάνο. Είναι ένα πρόβλημα η στη χώρα μου και υπάρχουν ορισμένοι δικαστές στην Ιταλία οι οποίοι πολλές φορές ασχολούνται με αυτά τα οποία κάνουν οι πολιτικοί και πάρα πολύ συχνά οι δικαστές αυτοί βρίσκονται χωρίς αρμοδιότητες, υφίστανται δυσμενείς μεταφέσεις κτλ. Συνεπώς λοιπόν το θέμα της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα το θέμα της δικαιοσύνης στην Ιταλία πρέπει να σας απασχολήσει. Θυμίζω ότι η Ιταλία έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για προβλήματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Θα ήθελα και τη θέση της Σουηδίας σχετικά με αυτά τα οποία είπε ο Μπερλουσκόνη χθε, σύμφωνα με το οποίο οι ε, εκπρόσωποι τύπου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να αναφέρονται σε θέματα δικαιοσύνης και σε θέματα εφαρμογής του νόμου στις διάφορες χώρες. Κυρία Παπαδοπούλου. Κυρία Υπουργέ, πράγματι είναι μεγάλο επίβολο το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι ξεκάθαρε οι δράσει και οι προτεραιότητε σα. Η συνεργασία τη χώρα μου, τη Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεδομένη. Εμεί θα συνεργαστούμε μαζί σα γιατί είμαστε το νοτιότερο σύνορο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το φλέγον πρόβλημα τη λαθρομετανάστευση από τρίτε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μα απασχολεί. Όμω το ερώτημα μου είναι ξεκάθαρο. Τι γίνεται με το 37% των κυπριακών εδαφών που είναι ευρωπαϊκά εδάφη και τελούν κάτω από τουρκική κατοχή τα τελευταία 35 χρόνια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στις κατεχόμενες περιοχές υπάρχει μια ανοιχτή πληγή, υπάρχει μια ανοιχτή τρύπα, υπάρχει λαθρομετανάστευση, υπάρχει παράνομος επικισμός, υπάρχει σωματεμπορία γυναικών και σωματεμπορία παιδιών, υπάρχει παράνομη δράση εγκληματικών στοιχείων δεν εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό Ένταγμα Σύλληψης και υπάρχουν ξεκάθαρα ονόματα, τα οποία γνωρίζομαι. Υπάρχει παραοικονομία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματο και όλα αυτά είναι ανοιχτέ πληγές για την Ευρώπη. Το ερώτημα μου είναι, τι σκοπεύει να κάνει η Σουηδική Προεδρία ώστε να προστατευτούν τα κατεχόμενα ευρωπαϊκά εδάφη της Κύπρου από τέτοια εγκλήματα και τι θα πράξετε για να πιεστεί η κατοχική Τουρκία τώρα που στο τέλος του χρόνου, το Δεκέμβριο του 2009, χτυπά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να έχει συμμορφωθεί προς τις διεθνείς της υποχρεώσεις. Η Κυπριακή επίσημη δημοκρατία, η επίσημη Κυπριακή Δημοκρατία θέλει ενδυνάμωση της Ευρωπόλ και όλων των διεθνών οργανισμών και ζητούμε τη βοήθειά σας για να προστατεύσουμε τα κατεχόμενα ευρωπαϊκά εδάφη της Κύπρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι διότι ως ε, νέα Ευρωβουλευτής μπόρεσα να ακούσω την Υπουργό μου είναι πολύ συγκινητικό αυτό για μένα και πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα το πολύ σημαντικό είναι η καταπολέμηση του εγκλήματος με τις ε, άπειρες μορφές που έχει αυτό. Κυρία Υπουργέ, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε όλες τις μορφές εγκλήματος και όντως πρόκειται για παραβίαση των ε, δικαιωμάτων μας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, εφαρμόζεται η νομοθεσία, προς ε, μεταφέρεται το κοινοτικό δίκαιο σε κάθε χώρα και θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν ελάχιστα ε, κριτήρια, μινιμουμ κριτήρια, τα οποία θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε παντού, ώστε να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα αδικαιώματα παρά το γεγονό ότι υπάρχουν διαφορέ ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Κυρία Μπορσελίνο. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα τα του οργανωμένου εγκλήματος, τα της τρομοκρατίας. Δεν άκουσα όμως να μιλάτε για τη μαφία, το οργανωμένο μαφιόζικο έγκλημα που είναι σχετικά διαφορετικό θέμα από άλλες μορφές εγκληματικότητας και απαιτεί διαφορετικά μέσα. Είναι προφανές ότι η ενίσχυση της Ευρωπόλ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όσοι έχουν ασχοληθεί με, την, με το οργανωμένο μαφιόζικο έγκλημα έχουν ε, δει τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν λόγω της έλλειψης επικοινωνίας και πληροφόρησης με άλλες χώρες γιατί πραγματικά η μαφία με τις πολλαπλές της μορφές έχουν ξεπεράσει τα σύνορα. Ε, θα ήθελα να μου πείτε τι θα πρέπει να κάνει η Σουηδική Προεδρία, τι σκοπεύει να κάνει η Σουηδική Προεδρία για την κατάσχεση των αγαθών της μαφίας και την ε, χρήση τους εκ των υστέρων. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες χρηματικές ποσότητες που δεν χρησιμοποιούνται. Στην Ιταλία υπάρχει ένας νόμος που επιτρέπει την κοινωνική χρήση των ποσών αυτών αλλά θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες, γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα επίσης ε, να δω τι γίνεται και με τους ε, προστατευόμενους μάρτυρες ε, στα πλαίσια της, των δικαστικών διαδικασιών εναντίον της μαφίας. Ξέρετε ότι λόγω ακριβώς της επικινδυνότητας των μαρτυριών τους ε, προστατεύονται με ειδικό τρόπο στη χώρα μου. Τι γίνεται ακριβώς και τι προβλέπει η Σουηδική Προεδρία γύρω από τα θέματα αυτά. Κυρία Χάνκης, τελευταία. Igen, örömteli volt és megnyugtató hallani miniszter asszony igazán kiváló és gondolatgazdag Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Υπουργό η οποία τόνισε πόσο σημαντική είναι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το οργανωμένο έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα, είναι διεθνές και η καταπολέμησή του απαιτεί να υπάρχει σε διεθνές επίπεδο συντονισμός. Όπως λοιπόν ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι, θα πρέπει να ενισχυθεί να διοριστή ο ρόλος της Ευρωπόλ. Η κυρία υπουργό ανέφερε πολύ σημαντικά θέματα και ανέφερε επίσης και τον συντονισμό. Μόνο κάποια στιγμή αισθάνθηκα όμως ότι υπάρχει μια κάποια αδυναμία. Γι' αυτό θα ήθελα να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, κυρία Υπουργέ. Πρόκειται για τις ε, οικονομικές ε, ε, συναλλαγές των τραπεζών offshore και την ε, σχέση τους με το οργανωμένο έγκλημα. Πώς μπορούμε να καταπαλεμήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο το φαινόμενο αυτό. Πολλοί το ανέφεραν το θέμα αυτό, το οικονομικό, με τους ε, τρομοκράτες και τις δραστηριότητες τους, αλλά θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί με ενδιαφέρει το θέμα αυτό όλος ιδιαίτερος. Η πατρίδα μου, η Ουγγαρία, πέρασε από το κομμουνιστικό καθεστώς σε δημοκρατικό καθεστώς σήμερα, αλλά πάρα πολλά πράγματα πρέπει να τα βελτιώσουμε ακόμη στη χώρα μας το οργανωμένο έγκλημα έχει μια κάπως ιδιάζουσα μορφή στην ε, Ουγγαρία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το θέμα αυτό και εγώ ως ε, διευθύντρια ενός Ινστιτούτου που ασχολείται με τέτοιου θέματα πρέπει να αντιμετωπίσω όλα αυτά τα θέματα αλλά αισθάνομαι κάπως αδύναμη. Περί τίνος πρόκειται. Όταν η Ουγγαρία και υποθέτω και άλλες χώρες που πέρασαν με ειρηνικό τρόπο από κομμουνιστικά καθεστώτα στα δημοκρατικά αντιμετώπισαν τέτοιου είδους θέματα όπου οι μυστικές υπηρεσίες και τα απομεινάρια τους κατά κάποιο τρόπο τα πρώτα λεπτά ήδη της αλλαγής της κατάστασης είχαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπολείπους είχαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπόρεσαν να μεταφέρουν σε τράπεζες του... Και έτσι δημιουργήθηκε ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος με πρώτους ε, εποφελούμενους, αν θέλετε, ε, πρώην ε, άτομα που συμμετείχαν στις ε, μυστικές υπηρεσίες και δημιούργησαν κάποιες ε, εταιρείε, κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ε, σχέση ακόμη με κάποια άτομα του προηγούμενου καθεστώτος που είχαν σχέση με τις μυστικές υπηρεσίες. Ναι, ναι, τελειώνω. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα ώστε να υπάρχει διαφάνεια και καλύτερη συνεργασία σε τέτοιου είδου θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο η Υπουργό σε πολύ λίγα λεπτά που έχουμε στη διαθεσή μας να απαντήσει. Είμαι σίγουρος όμω ότι θα το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, για τα σχόλια που υποβάλατε και τις δεσμεύσεις που αναλάβετε σε κάποια θέματα. Αυτό είναι θέμα εμπιστοσύνης των πολιτών και προς τα θεσμικά όργανα και ενδιαφέρει όλους τους πολίτες να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό όμως που τους απασχολεί επίσης είναι πώς θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε αποτελεσματικά μέτρα και πώς θα τα εφαρμόσουμε για να φέρουμε σε πέρα σε αυτή την ε, αποστολή μας. Έχουμε μπροστά μας πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά τους επόμενους μήνες. Θα ήθελα απαντώντας να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι εκφράστηκαν κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης της, ε, της ε, νομοθεσίας ε, είναι αποτελεσματικός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε εμείς το οργανωμένο έγκλημα και πώς γίνεται η αξιολόγηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη αξιολόγηση, καλύτερη εκτίμηση της νομοθεσίας και να πούμε τι ακριβώς ξέρουμε, πού μπορούμε να, και δεν ξέρουμε καλά, πού μπορούμε να βελτιωθούμε ώστε τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε να είναι εύστοχα και αποδοτικά. Ένας βουλευτής ε, από την ομάδα των Πρασίνων είπε ότι θα πρέπει πριν να υιοθετήσουμε νέα μέτρα, κάνουμε αξιολόγηση των μέτρων των οποίων έχουμε τώρα στη θέση μας και εφαρμόζουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι μια αξιολόγηση από πολιτική σκοπιάς. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι ε, προχωρώντας και έχοντας καλύτερη εμπειρία να εφαρμόζουμε τα μέτρα Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να εφαρμόζουμε μέτρα και κάνουμε μόνο αξιολόγηση του παρελθόντος. Και νομίζω ότι ε, αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Τώρα, στα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στα PNR των επιβατών χρησιμοποιούνται και για να αυξηθεί η ασφάλεια των ε, ε, επιβατών και στο αεροδρόμιο της Ατλάντα χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε Πώς θα χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία ξεκινώντας από ποιο σημείο αναφοράς, ε, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε και ποια είναι τα κριτήρια που θα εφαρμόσουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Εάν χρησιμοποιούνται σωστά τα δεδομένα, αναμφίβολα μπορούμε να Θα αξιοποιήσουμε σωστά, λαμβάνοντας υπόψη ποιε είναι οι δομές που διαθέτουμε και ποιοι είναι οι κώδικοι, συγγνώμη, που θα ακολουθήσουμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είναι εύκολο το θέμα, το καταλαβαίνω. Επίσης έγιναν πολλές ερωτήσεις για το SWIFT και την ανταλλαγή δεδομένων. Πρέπει να πω ότι θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για τέτοιου είδους θέματα. Και εμείς ε, εκ μέρους της Προεδρίας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να βελτιωθεί η συνεργασία μας. Η ορατότητα του τι ακριβώς κάνουμε και η διαφάνεια είναι σημαντικό για μας. Δεν θα πρέπει να είμαστε αρνητικοί. Επίσης, πρέπει να πω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να, έχουμε, ε, να μπορούμε να εγγυηθούμε την ακαιρεότητα των δεδομένων. Βεβαίως, σε όλες τις ε, συζητήσεις θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εμείς εκ μέρους του μας Προεδρίας κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ανοίξουν τα στοιχεία, να ανοίξουν οι φάκελοι. Ό,τι πληροφορίες έχουμε βεβαίως μπορούμε να τις μεταφέρουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην έχετε την εντύπωση ότι εμείς δεν θέλουμε να σας ενημερώνουμε. Θέλουμε ε, όλα τα μέσα που διαθέτουμε, όλες τις πηγές πληροφοριών να τις αξιοποιήσουμε σωστά και βεβαίως ό,τι στοιχεία έχουμε, θα σας τα διαβάζουμε. Τώρα, η καταπολέμηση της μάφιας, του οικονομικού εγκλήματος, του οργανωμένου εγκλήματος, ε, για να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, έχουμε πολλά μέσα στη διαθεσή μας, αλλά σίγουρα χρειάζεται βελτίωση. Και σίγουρα θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αξιολογήσουμε περισσότερο διάφορες πηγές πληροφοριών που έχουμε πολλές φορές ε, ε, οδηγεί στην εγκληματικότητα το χρήμα, τα οικονομικά συμφέροντα. Και αν ε, αρχίσουμε καταπολεμώντας αυτή την πτυχή του προβλήματος, τα οικονομικά συμφέροντα σίγουρα θα έχουμε και στην καταπολέμηση του γραμμένου εγκλήματος καλύτερη αντιμετώπιση. Διότι Έτσι θα προλάβουμε και περαιτέρω αύξηση τέτοιου είδους ε, ε, εγκληματών. Η κυρία, ε, μία συνάδελφό σας, μίλησε για θέματα ασυμβατότητας και μεταξύ δύο αποφάσεων πλαισίου. Κάποια στιγμή υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία, αλλά κάποια στιγμή υπάρχουν και επικαλύψεις μεταξύ των αποφάσεων που έχουμε. Πολλές φορές ε, υπάρχουν ε, πληροφορίες οι οποίες αφορούν ε, κάποιες περιπτώσεις εγκληματικότητες οι οποίες είναι κατακαιρματισμένες αναχώρα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε εμείς να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες ώστε να έχουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για να καταπολεμήσουμε καλύτερα το οργανωμένο έγκλημα. Διαφορετικά, ένα γενικότερα ε, σημασίας ε, θέμα μπορεί να κατακαιρματιστεί, να υπάρχουν πληροφορίες δηλαδή ε, πιο κατακαιρματισμένες και να μην μπορεί κανείς στη να δει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση για να το επιλύσει πιο εύκολα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα προετοιμαζόμαστε κάθε φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων που μας απασχολούν. Πρέπει να πω ότι σε θέματα επίσης ε, διαδικαστικά φαίνεται ότι κάποιοι πιστεύουν ότι δεν έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Τόσα, όσον αφορά το δικαίωμα των ε, κατηγορούμενων για διάφορα ε, παραπτώματα για δικήματα να καταλαβαίνουν στη γλώσσα τους γιατί κατηγορούνται για να μπορέσουν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ε, ενδεχομένως κατηγορουμένων. Κάθε χώρα ξέρουμε ότι έχει διαφορετικό σύστημα και τα συστήματα, το σύστημα κάθε κράτους έχει διαφορετική δομή και ξέρουμε ότι κάποιος όταν κατηγορείται, ε, θα πρέπει όμως να δυσκολεύσουμε ότι αν κάποιος κατηγορείται για κάποια πράξη σε μια άλλη χώρα που δεν είναι η δική του, να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται και ποια είναι τα δικαιώματα που έχει για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δεδομένου ότι αυτό είναι από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα του ανθρώπου. Όλοι ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ένα από τα κυρίαρχα δικαιώματα είναι η ελευθερία της έκφρασης. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς θα μπορούμε εμείς στα πλαίσια της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης των πολιτών μας να ενεργήσουμε στον τομέα της δικαιοσύνη χωρίς να καταστρατηγούμε αυτό το δικαίωμα και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες να ε, ξεπεράσουμε τέτοιες δυσκολίες. Μακρηγορώ, λέει η Υπουργό. Τώρα, Όσον αφορά την Ευρωπόλ, συμμερίζομαι τις ε, απόψεις σας. Όντως μπορεί να βελτιώσει το προφίλ της, ε, το θετικό, να βελτιώσει το ρόλο της και το έργο της η Ευρωπόλ. Και πιστεύω ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Βένράιτ, ο πρόεδρος της Ευρωπόλ, όταν ε, ε, ρωτάτε η Ευρωπόλ, έχετε αρκετούς πόρους για να ενεργήσετε, έχετε αρμοδιότητες επιχειρησιακές για να ενεργήσετε. Η Ευρωπόλ θα πρέπει να είναι σε θέση, εκτός των άλλων, να κάνει και συντονιστικό έργο στα πλαίσια των καθηκόντων που τις έχουν αναθέσει οι διάφορες ε, αρχές των κρατών μελών, για να είναι πιο αποτελεσματικό. Εγώ συμμερίζομαι αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος του Ευρωπόλου, ο κ. Ράιτ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να μπορεί κανείς να αποδείξει ότι μπορεί να συντονίσει για να προσφέρει αυτή την υπεραξία, αυτό το συν. Δηλαδή, να κάνει κάτι περισσότερο από ό,τι μπορεί να κάνει κάθε αρχή σε εθνικό επίπεδο. Τελειώνοντα, θα ήθελα να σα πω ότι ούτω ή άλλω είμαι στη διαδικασία και εγώ και οι συνάδελφοι υπουργοί για να επανέλθουμε και να εξηγήσουμε οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλετε να μα θέσετε. Πρέπει να σα πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ τι ερωτήσει σα. Κατά τη διάρκεια όλη τη Προεδρία μπορείτε να μα απευθύνετε Οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί, ε, θέλετε μέσω email και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε, μπορούμε κάθε φορά να απαντούμε στα ερωτήματά, μας, στα ερωτήματά σας. Συγγνώμη. Και ελπίζω ότι όλοι ενωμένοι θα βοηθήσουμε προς την καλύτερη ε, και αποτελεσματικότερη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και όποιας μορφής τρομακτικής. Ευχαριστώ πολύ. Minister, Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ, για την εξαιρετική σας δουλειά. Σας ευχαριστούμε για τον καρποφόρο διάλογο στον οποίο μας οδηγήσατε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Όπως είπε η υπουργό, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τομπίας Τίλστρομ, θα είναι το απόγευμα μαζί μας στις 3. Ξέρετε ότι στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης και ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί αμέσως τώρα σχετικά με τη γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό για το 2010. Αλλά έχουμε ήδη ξεπεράσει το χρόνο τώρα. Γι' αυτό προτείνω να ε, κηρύξουμε τη λήξη εδώ της πρωινής συνεδρίασης και να αναβάλουμε τη συζήτηση για τον προπολογισμό αμέσως μετά την ε, παρουσίαση του κυρίου ε, Μπίλστρομ το απόγευμα. Και αμέσως μετά από αυτήν θα ε, σκεφτούμε, θα συζητήσουμε δηλαδή τα θέματα του προπολογισμού. Αν συμφωνείτε, στις 3 λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Α, κυρία Μπόσκουρτ. Ένα μικρό διαδικαστικό Έχουμε τώρα μεν την Σουηδική Προεδρία, αλλά ποτέ δεν είχαμε ε, από τη Γαλλική Προεδρία ή την Τσεχική Προεδρία τον αρμόδιο υπουργό για την οδηγία εδώ. Ίσως ο υπουργό Σαπούνη είναι αρμόδιος, θα μπορούσε να προσέλθει ενώπιόν μας και να απαντήσει σε ερωτήσεις. ο πρόεδρος. Το σημειώνουμε αυτό. Στις 3 λοιπόν, τον Πίας Φίλστρομ. See you, see you tomorrow. Yeah, I didn't introduce myself. Tomasz Bańka.